Έχουν ήδη περάσει 6 λεπτά μετά τις 9. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε αρκετά υπερφορτωμένη την ημερήσια διάταξη με τις ψηφοφορίες, οπότε θα σας παρακαλούσα χωρίς άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες που προβλέπετε να διαρκέσουν για καμία ώρα περίπου. Σημείο 17. Ε, προπολογισμό, απαλλαγή για το 2017, Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Είναι η Ναγκίλ, είναι η συγγετριά μα. Απουσιάζει όμω. Οπότε, αν δεν θέλει άλλο συνάδελφο το λόγο, να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αλλά ας το ελέγξουμε καλό κακού. Για προθέρμανση κιόλα. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 20. Τέλος. Απορρίπτεται τελικά. 21. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. ...52 είναι παρόντες, 51 έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία και με 44 ψήφους υπέρ 6 ε, κατά εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Οπότε περνάμε στο 18 απαλλαγή 2017, ε, Γενικός Προϋπολογισμός και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η και πάλι συντάκτρια γνωμοδότηση. Αν δεν θέλει κανείς το λόγο να περάσουμε στην ψηφοφορία. ξεκινώντα από την τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ποιο είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχέ. απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά απόχέ. ηλεκτρονικός έλεγχος για το 18 άρχεται η ψηφοφορία. Ε, με μικρή διαφορά απορρίπτεται. Αυτή ήταν η 18. Πάμε στη 19 του κυρίου Πρέντα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και 20 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σχέδιο γνωμοδότης. Άρχεται η ψηφοφορία. Δύο δεν ψήφισαν. Ένας. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 41 ψήφους υπέρ και 3 κατά. Επόμενο σημείο, 19. Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών του αφενό και τη Αραβική Δημοκρατία τη Αιγύπτου αφετέρου για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση τη Δημοκρατία τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκίτρια είναι η κυρία Μανέσκου που απουσιάζει. Μπορούμε όμως να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο σύστασης. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 48 υπέρ και μία ψηφοκατά. κατά. Επόμενο σημείο, Συμφωνία Συνεργασία για την Εταιρική Σχέση και την Ανάπτυξη μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ισλαμική Δημοκρατία του Αφγανιστάν. Θέμα που συζητήσαμε χθε το απόγευμα. Η η ε, κυρία Φωτίκα κολλείεται. Ο κύριος Στάνοκ την αντικαθιστά, δεν ξέρω θέλει να σχολιάσει κάτι. Όχι, οπότε περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία που θα γίνει ηλεκτρονικά, άρχιτη ψηφοφορία.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 δεν με είχαν ενημερώσει, έχουμε μία ηλεκτρονική ψηφοφορία, αυτό μου λέει η γραμματεία, για τη συγκατάθεση, τη συνένεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πείτε παρακαλώ ότι ψηφίζουμε στους συναδέλφους. Ψηφίζουμε πρώτα την συνένεση και μετά το ψήφισμα που τη συνοδεύει. Μπορούμε επιτέλους να ξεκινήσουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Δεν ψήφισαν όλοι. Εσείς δεν ψηφίσατε. Τέλος, 45 υπέρ, 3 κατά. τώρα θα περάσουμε στο 21, το ψήφισμα δηλαδή για το Αφγανιστάν. Δεν υπάρχουν σχόλια, ψηφίζουμε το ψήφισμα για το Αφγανιστάν. Συμβαστική τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Λυπάμαι μικρό λάθος. 69 τροπολογία πρώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικό ηλεκτρονικός έλεγχος για την 70, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται. η 71 και 72 καταπίπτουν. Πάμε στην 74. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 74, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 75. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά αποχές. 76. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 78. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 88. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 101. Δεύτερο τμήμα μόνο. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100 Κατά τμήματα θα ψηφίσουμε. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα, άρχιτη ψηφοφορία. It's Τέλος, με μικρή διαφορά εγκρίνεται οριακά. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 120? Ευχαρίστω. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 120. It's been adopted. 121. Εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 121. άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και αυτή. 134 υπέρ κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 134, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 137, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται με διαφορά. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 125 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος και απορρίπτεται. 126. Ποιος είναι υπέρ της κυρίας Λέζικ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125 απορρίφθηκε και γι' αυτό χρειάστηκε να ψηφίσουμε και την 126 που κατα... απορρίφθηκε και αυτή και πάμε στην 127 του κυρίου Σαφοζέρ. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. Oh. Δεν Και 128 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Καταπίπτει η 227, 144 υπέρ κατά. Αποχές επαληθεύουμε παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. 14 συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά εγκρίνεται. 153 συγγνώμη. 119 κατά Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έτσι δεν είναι. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΔΕΒΕ 8 υπέρ Κατά. Δεν έχει καταπέσει. Θα σας παρακαλώ μην επεμβαίνετε. Δεύε 8 υπέρ κατά αποχές. Δεν συμμετέχει και κανείς. Εγκρίνεται. 18 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 173 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε. Καλώς, να το πάω πιο αργά, κανένα πρόβλημα. DV1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν εγκρίνεται, μάλιστα. Ε, πέντε της ΔΕΒΕ υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεβετρία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά αποχές Δεβε ΔΒ10 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε τη 10 της ΔΕΒΕ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται του κυρίου Φρουντζούλητσα καταπίπτει δεν πέφτει ο ίδιος η τροπολογία του καταπίπτει 192 losing υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 193 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί επαληθεύουμε 193 Πέρας. Απερίφθη. 194 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. <laughs> Πιο πολλές είναι παρά οι πέτρες στην έρημο του Αφγανιστάν, λέει ο πρόεδρος. 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ Πέρας. Εγκρίνεται 201 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί. 202 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί. 203 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 204 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 205 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 206 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 207 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 208 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται μάλλον. να δούμε τι κάνει άλλη. Καλά, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 208. Επαλήθευση. πέρας εγκρίνεται 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η ΤΕΒ 7 καταπίπτει 213 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε τη 213 αρχής ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται 2.14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.17 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε 217 Πέρας εγκρίνεται 218 υπέρ κατά αποχές Επαληθεύουμε και τη 218, αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 219 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ. Κατά αποχές. Αμέλ. Επαλήθευση. 221. Πέρας. Εγκρίνεται. 222 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 224 υπέρ κατά αποχές. Επαληθεύουμε τη 224 αρχής ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 225 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 226 υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε τη 226, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 228 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 55 καταπίπτει. 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τη 229 θα ελέγξουμε. Μάλιστα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Προφανώς εγκρίνεται. 24 συμβαστική υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές Ας αλλάξουμε και την 9 παρακαλώ. Αρχίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές. Επαληθεύουμε τη 10. Πέρας. Εγκρίνεται. Σαφές. 12 υπέρ κατά αποχές. Απεριφθεί. 13 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ καταπίπτει. Και πάμε στη συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 βαλέρο υπέρ κατά αποχές. Λοιπόν, ας κλείσουμε το 21, έχει εγκριθεί έτσι και ζητήσατε την 22-25 on block. Όχι, αδύνατον λοιπόν.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 αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε τη 43 αρχής ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογικές αναφορές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε την 5 της κυρίας Βαλέρο. Πέρας. Εγκρίνεται. 28 υπέρ, 26 κατά. Υπαριθμόν 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και το σύνολο για ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σχέδιο εκθέσεως όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 50 υπέρ, 3 κατά. Και τώρα σημείο 22. Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμφωνία της και Δημοκρατία τη Σιγκαπούρη. Ο κύριο Αντώνιο Λόπε Ιστούρη Χουάιτ. Αν θέλετε να πείτε κάτι, κύριε συνάδελφε, όχι. Και ψηφίζουμε. Ενημερώνω για άλλη μια φορά πω πρώτα κάνουμε με μία ψηφοφορία την χορήγηση τη συνένεση. ηλεκτρονικά παρακαλώ, αρχίζει. Τη σύμφωνη γνώμη, συγγνώμη. Πέρας και έγκρινεται. 50 υπέρ, 3 κατά, 4 εποχές. Ψήφισμα. Για την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τι ενάμει συμφωνίε εταιρική σχέσει και με μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία Σιγκαπούρη. Ρωτώ και πάλι τον εισηγητή αν θέλει κάτι να πει. Ιδάλω περνώ στην ψηφοφορία. Ξεκινώ με τη 16 κύριε, του κυρίου Μπίτικοφερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά, συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά Επαληθεύουμε την 24 παρακαλώ, αν αρχίσει η ψηφοφορία. Λείπουν δύο ψήφοι. Πέρας. Εγκρίνεται 29 υπέρ, 25 κατά. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρκατα κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρκατα κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρκατα κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 47 υπέρ κατά αποχές απερίφθη έτσι. 47 λοιπόν, έχει απορρίφθει 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, αιτιολογικές σκέψεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ κατά κατά αποχές απερίφθη 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την 8 Πέρας και εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκατέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απερίφθη συγγνώμη, 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τιολογικές αναφορές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ηλεκτρονικά περνούμε στο ε, σύνολο, όπως τροποποιήθηκε το ψήφισμα παρακαλώ. Πέρας. Και εγκρίνεται. 49 υπέρ, 2 κατά, 6 εποχές. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο 24. Έτσι λοιπόν έχουμε την έκθεση του ΕΚ σχετικά με την στρατηγική επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους δύο έτη μετά από την έγκρισή της. Η κυρία Φωτίγκα, η συγγήτρια, δεν είναι μαζί μας σήμερα για τη σύσταση αυτή προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και είπατε εκπρόσωπο της Ένωσης. Άρα λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιο θέλει να πει δύο λόγια εκ μέρους της. Εάν όχι, θέλω να τα δούμε ένα-ένα από το κατάλογο ψηφοφοριών. Αμάλ, κάτι έχεις να πεις? Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ, Δεν υπάρχει 63. Έχουμε τον παλιό κατάλογο μάλιστα. Λοιπόν, πού ήμουνα, ήμουνα στο 63, λυπάμαι πολύ Ραμόνα, δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Ραμόνα Μονέσκου, η τροπολογία σου, υπέρ, κατά, αποχές, υπέρ, είναι η πλειοψηφία, 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 65 υπέρ, κατά, αποχές. Για να δούμε την 65 ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 του κυρίου Καστάλντο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 στην 185 ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Λυπάμαι, αγαπητέ συνάδελφε. Ε, την συμβαστική 18 την ψηφίσαμε. Και τη 19 την ψηφίσαμε και τώρα περνάμε προς γενικότερη έκπληξη. Θα περάσουμε λοιπόν στη συμβιβαστική 20. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 215 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ το 215. Υπέρ, ε, άρχεται η ψηφοφορία, με συγχωρείτε. Πέρας. Απορρίπτεται. 216 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 231 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.46 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 258 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 259 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 260 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 261 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 262 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν σε εκτιμώντας. Συμβιαστική υπορθμόν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα περάσουμε τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία για το σύνολο της ε, έκθεσης ως τροποποιήθηκε. Πέρας εγκρίνεται 49 επέρ 7 κατά. Δύο εποχές. Θα ήθελα να σας συγχαρώ. Μπορούμε τώρα λοιπόν να περάσουμε στην εφαρμογή του κανονισμού σήμα ΓΑΜΑΠΗ ε, αριθμός 978 του 2013. Εισηγητής ο κύριος Παντζέρη. Θέλετε να πάρετε το λόγο? Όχι. Μπορούμε λοιπόν αμέσως να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατα, κατά αποχές θα ήθελα ηλεκτρονικά τη συμβιβαστική υπαριθμό 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 38-2. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές. Την 27 παρακαλώ ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά την 34 παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικά την 41 παρακαλώ, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ ηλεκτρονικά τη 42 παρακαλώ. Πιστεύω πως ε, αλλά θέλω να το δούμε και ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά και τη 45 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασ... Με συγχωρείτε, η 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικά την 56 γιατί είχα πάρα πολλές αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε συμβαστική ενέα λοιπόν. Υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικά την συμβιβαστική ενέα Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίθηκε. 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σε αιτιολογικές σκέψεις η πρώτη υπέρ. Κατά αποχές την υπαριθμόν να παρακαλώ ηλεκτρονικά άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Υπάρχουν 2, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικά και εδώ, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας, απορρίπτεται. Η 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 4, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικά παρακαλώ και υπαριθμό 4 εδώ, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7. Urban Crespo υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά και την υπαριθμόν 7. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σχέδιο γνωμοδότησης ως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται 50 υπέρ, 2 κατά, 6 αποχές. Σας είχα υποσχεθεί στις 10, είναι 7, είναι 10 παρά 7. Έχουμε λοιπόν και 7 λεπτά στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. So, colleagues, let's... Συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Μετά από μία ώρα ψηφοφοριών, περνάμε στο σημείο 26, την ενημέρωση σχετικά με την αποστολή της Επιτροπής μας στο Ιράκ και το Ομάν, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Περάσαμε δύο μέρες στη Βαγδάτη και δύο μέρες στο Μουσκάτ. Η ενημέρωση θα γίνει παρουσία του επικεφαλής αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ, του κυρίου Ραμόν Μπλεκούα, τον οποίο καλωσορίζω θερμότατα. Έτυχε να βρίσκεται στις Βρυξέλλες σήμερα και θα του δώσω το λόγο για μια σύντομη παρέμβαση σε λίγο. Ε, θα ήθελα επ' ευκαιρία να σας ευχαριστήσω κύριε Πρέσβη για την οργάνωση της επίσκεψής μας στη Βαγδάτη που ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, επίκαιρη και μείζωνος πολιτικής σημασίας. Εμείς η αντιπροσωπεία της ΑΦΕΤ είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε πολύ σημαντικές συζητήσεις με ηγεσία του Ιράκ στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Μεταξύ άλλων συναντήσαμε τον πρόεδρο του Ιράκ, τον πρωθυπουργό, τον υπουργό εξωτερικών και τον αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράκ. Στις περισσότερες συναντήσεις μας οι συνομιλητέ μας, οι Ιρακινοί μα ενημέρωσαν για την πρόθεσή τους να απαλλαγούν από ανάμειξη των ξένων στις εσωτερικέ του υποθέσεις και διατρένωσε το στόχο του Ιράκ να γίνει μια θετική γέφυρα μεταξύ των περιφερειακών δυνάμεων. Είμαι σίγουρη, σίγουρος ότι η επίσκεψη αυτή συνέβαλε στην ενίσχυση της πολιτικής διάστασης της συνεργασίες, ε, Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράκ και με αυτή την άποψη πιστεύω ότι θα συμβάλλουμε στο να υλοποιήσει, ε, προσβλέπω μάλλον και ελπίζουμε να πραγματοποιήσει όλο το Ιράκ την πολιτική, οικονομική και κοινωνική του σταθερότητα. Και στο Μάν ήταν επιτυχής η επίσκεψή μα, Συναντηθήκαμε με τους Προέδρους του Συμβουλίου της ΣΟΥΡΑ και του Συμβουλίου του Κράτους και τον ε, Υπουργό Εξωτερικών Μα ενημέρωσαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντο, όπω η κρίση στο Συμβούλιο του Συνεργασία του Κόλπου, τι ε, συγκρούσει στην Ιεμένη, Συρία, Λιβύη και την εθνική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, καθώ και τα σχέδια του Ιράν να διαφοροποιήσει την οικονομία του και να μειώσει την εξάρτησή του από του υδρογονάνθρακε. Ε, Τέλο, συνειδητοποίησαμε πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο του ΟΜΑΝ ε, ω διαμεσολαβητή σε πολλέ τοπικέ συγκρούσει. Αυτά ε, εισαγωγικά. Θα δώσω το λόγο στον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ, τον κύριο Ραμόν Πλεκούα και μετά αν το επιθυμεί στην κυρία Μισελ Αλιό Μαρή που είναι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τη σχέση μας με την Αραβική Χερσόνησο. Θα ακολουθεί η συζήτηση. Κύριε Μπλεκού, έχετε το λόγο, κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσω μαζί σας ε, στο πλαίσιο του Ιράκ το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι έγινε σε πολύ κρίσιμη στιγμή αυτή η αποστολή της ΑΦΕΤ, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ιράκ. Γιατί βρισκόμαστε στην έναρξη ενός νέου πολιτικού κύκλου στο Ιράκ. Και όπως θα διαπιστώσετε από τις συζητήσεις που είχατε με όλους τους πολιτικούς ηγέτες ε, των δύο βασικών συνασπισμών, έχει αλλάξει το αφήγημα δεν μιλούν πλέον για ε, εθνοτικές συγκρούσεις ή ε, την ε, διαμάχη για τη διεκδίκηση ισχύω, αλλά περάσαμε σε νέο αφήγημα για την παρασυμφιλίωση, την ενοικοδόμηση και τη συνεργασία την διεθνωτική. Και μετά την δύσκολη πολιτική κρίση που πέρασε πέρυσι το Ιράκ, είδαμε επιτέλους μία ειρηνική μετα... μεταβίβαση ε, ισχύω. Και αυτή είναι απόδειξη της ελληνικής Δημοκρατίας. Μπορεί να έχει ελλείψεις και αδυναμίες και πολλές προκλήσεις, αλλά είναι το συμπεφωνημένο πλαίσιο στο οποίο οι διάφοροι πολιτικοί ε, παράγοντες μπορούν να καταλήξουν συμφωνία. Και αυτό πραγματικά είναι ιδιαίτερη περίπτωση στην περιοχή, κάτι εξαιρετικό δίνει λόγο ικανοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμβολή της, τη συνεισφορά της στη διαδικασία αυτή. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι η όλο και μεγαλύτερη εμφάνιση διεθνώς του Ιράκ. Και μετά την ε, ανάδειξη της νέας κυβέρνησης 24 Οκτωβρίου, Είχαμε έναν οργασμό διπλωματικών δραστηριοτήτων. Ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός και ο νέος υπουργός εξωτερικών συνεργάζονται με ταχύτατους ρυθμούς και με πολλή συνεργασία μαζί με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και προσπαθούν να κάνουν διαβήματα προς ε, περιφερειακές δυνάμεις και χώρες και τους διεθνείς εταίρους προσπαθώντας να υπογραμμίσουν το νέο ρόλο που θέλει να διεκδικήσει και να διαδραματίσει το Ιράκ. Να μην είναι απλώς πεδίο μάχης μεταξύ αντιμαχόμενων πλευρών, αλλά να γίνει γέφυρα που θα συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα. Αυτές είναι οι βλέψεις του Ιράκ. Και όπως είπατε, το Ιράκ δεν θέλει να γίνει ένα εργαλείο σε αυτή την πάλι τη διαμάχη για την διεκδίκηση ισχύω, αλλά θέλει να γίνει γέφυρα μεταξύ των περιφερειακών γειτόνων της και των διεθνών εταίρων και ε, θέλει υποστήριξη για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο της γέφυρας. Και μάλιστα πρόσφατα, μετά την επίσκεψη του Πρόεδρου Τραμπ που έγινε σε ε, προσδόκητες και ειδικές συνθήκες, είχαμε και την ε, επίσκεψη του Υπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας και του Βασιλέως της Ιορδανίας και μάλιστα συνέπεσαν την ίδια μέρα όλες αυτές οι επισκέψεις. Είχαμε σαν το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες, ήταν άνευ προηγουμένου. Και πραγματικά εξήστε με πώς κατάφερε η Ιρακινή διπλωματία να χειριστεί τόσες πολλές επισκέψεις τόσο, τόσο υψηλού επίπεδου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πάντως τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, το Ιράν, και οι χώρες της περιοχής ε, και οι ευρωπαϊκές χώρες όλοι χρειάζονται το Ιράκ και θέλουν το Ιράκ να παραμείνει σταθερός και επικοδομητικός εταίρος στην ευρύτερη περιοχή. Και από αυτή την άποψη όλοι νιώσαμε και αυτό το αίτημα των, Ιρανι... Ιρακινών αρχών να ε, συνδέσουν την πολιτική τους ε, και να την αγκιστρώσουν στην πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι έπαιξε και συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο που συμβαδίζει με το αίτημα του Ιράκ να συνεχίσει να παίζει αυτό το ρόλο στην ε, ανοικοδόμηση των απελευθερωμένων ζωνών και στην διαμόρφωση της πολιτικής περιφερειακής σταθερότητας. Πέρυσι ξεκινήσαμε με την έγκριση της νέας στρατηγικής για το Ιράκ. Συνεχίζουμε με το ρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Πατή έπαιξε στη διάσκεψη του Κουβέιτ που συμπροέδρευσαν στην, στην διάσκεψη αυτή. Μετά εγκρίθηκε η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που θα αποτελέσει το πλαίσιο για μια πιο μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση. Και νομίζω ότι αυτά είναι τα εργαλεία που έχουμε, οι μηχανισμοί, μαζί με την δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ανοικοδόμηση, την ανασυγκρότηση του Ιράκ με σημαντικό κονδύλιο για τη συνεργασία που μας εφοδιάζει με όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε. Και θέλουμε και την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς, αυτά τα μέσα και να τα καταστήσουμε πιο επιτυχή και αποτελεσματικά για να υλοποιήσουμε και την παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πρωταρχικό της στόχο που είναι η συμβολή στην πρόληψη των συγκρούσεων και στη διευθέτηση των κρίσεων. Προκειμένου να επεκτείνουμε αυτή τη σφαίρα σταθερότητας και ευημερία ε, στην περιοχή μας, γιατί η σταθερότητα δεν ξεκινάει στα σύνορά μας. Η σταθερότητα ξεκινάει σε μια χώρα σαν το Ιράκ. Το Ισλαμικό κράτος ε, είναι απειλή για τις πόλεις μας, αλλά το Ισλαμικό κράτος ξεκίνησε από το Ιράκ. Από εκεί προέρχεται. Και πιστεύω ότι το Ιράκ ήταν ίσως το πιο επιτυχημένο μοντέλο για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και για την καταπολέμηση του ιδεολογικού νιχιλισμού, ε, μηδενισμού που εκπροσωπεί το Ισλαμικό κράτος. Γιατί το, το Ισλαμικό κράτος σε άλλες χώρες ε, ενεργοποιείται πολύ περισσότερο από ό,τι στο Ιράκ που εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Αλλά δεν είναι πια περιφερειακή δύναμη και σημαντική δύναμη. Βέβαια, είναι ένα αντάρτικο και η μάχη συνεχίζεται γιατί δεν έχει εξολοθερευτεί το Ισλαμικό κράτο. Αλλά εξακολουθούμε να στηρίζουμε την εθνική στρατηγική ασφαλεία του Ιράκ, την αντιτρομοκρατία, την, τον συντονισμό με τις, υπηρεσίες, τις μυστικές υπηρεσίες και μάλιστα είχαμε ε, μία συνάντηση ε, Συντονιστική Συντονιστική με έτοιμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει και να ενισχύσει αυτή την συμμετοχή της, την δέσμευσή της. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία ρηξικέλευθης μεταρρύθμισης των οικονομικών και πολιτικών δομών της χώρας. Το Ιράκ υπολογίζει σε μας και είναι ευγνώμων για τη συνεισφορά μας και τη δέσμευσή μας στη χώρα. Αν με ρωτάτε τώρα κατά πόσο η κυβέρνηση του Αμπτέλα Δελμάχτη θα έχει επιτυχία. Θα μπορούσα να σας δώσω ε, λόγους, γιατί θα μπορούσε να τα καταφέρει, αλλά και ποιες είναι οι επιλέσεις και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει. Οπότε δεν μπορώ να προβλέψω αν θα είναι επιτυχής ή όχι η διακυβέρνηση. Αυτό που μπορώ να σας προβλέψω είναι ότι το κόστος της αποτυχίας στο Ιράκ για τους ίδιους τους Ιρακινούς αλλά και για τη διεθνή κοινότητα θα είναι τεράστιο. Το τίμημα της αποτυχίας θα είναι τεράστιο γιατί το Ιράκ εξακολουθεί να είναι ως λίθος σταθερότητα στην περιοχή και είναι ένας παράγοντας, ένας φορέας, ένας παίκτη που μπορεί να έχει συνομιλήσει με όλες τις άλλες δυνάμεις. Μάλιστα σε μια στιγμή που η ένταση έχει αυξηθεί, έχει κλιμακωθεί. Οπότε είναι προς το συμφέρον μας να συμβάλλουμε στην υλοποίηση της επιτυχίας του Ιράκ. Και υπάρχουν στοιχεία που συμβάλλουν σε αυτή την ευόδοση των σχεδίων. Υπάρχει αποφασιστικότητα και βούληση της ηγεσία να βρεθεί πολιτική συμφωνία που θα επιτρέψει τη συνέχιση της πολιτικής διαδικασίας και την αποτροπή εσωτερικών διενέξεων και υπάρχει και η δεδηλωμένη πολιτική βούληση να παίξει το ρόλο της γέφυρας ε, το Ιράκ στην περιοχή. Και είναι προς το συμφέρον να στηρίξουμε αυτά τα σχέδια. Και η επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέβαλε ακριβώς στην διατράνωση αυτής της δέσμευσης, γιατί τα μηνύματα ήταν ξεκάθαρα και μάλιστα ε, έγιναν δεκτά με ικανοποίηση. Και σίγουρα έχουμε και τα μέσα να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα σχέδια και τα μηνύματα. Αυτά. Είναι μια ιδιαίτερα περίπλοκη και παράδοξη χώρα το Ιράκ. Σίγουρα θα έχετε απορίες και πολύ ευχαρίστω να απαντήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Πρέσβε για την σύνοψη που μας κάνατε, την κατατοπιστική για την κατάσταση στο Ιράκ. Αυτά διαπιστώσαμε κι εμείς το διήμερο που περάσαμε εκεί και, και εσείς και ο Βρετανός ε, πρέσβης φαντάζομαι ήταν πολύ άσχολοι δεδομένου με το μεγάλο αριθμό των διεθνών επισκέψεων. Θα δώσω αργότερα το λόγο στην κυρία Λιωμάρη, γιατί είναι αρμόδια μόνο για το ΟΜΑΝ. Ε, θα μιλήσουμε πρώτα για το Ιράκ, οπότε... Ρωτώ τους συναδέλφους αν θέλουν να περιοριστούμε σε αυτά που είδαμε στις δύο ημέρες της επίσκεψης στη, Μαγδα, στη Βαγδάτη, Ντονζόν, Γκόμες, Μπούχνερ, Κάρβα ο κύριος Νόμζον πρώτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόκειται για μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αποστολές που είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε στη διάρκεια αυτής της βουλευτικής περίοδου από την Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ τον πρέσβη, ευχαριστώ τη γραμματεία. Μπορέσαμε να συναντήσουμε αυτούς που πράγματι έπρεπε να συναντήσουμε, Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε μείνει και περισσότερο. Αισθανθήκαμε δυσφορία μόνο γιατί δεν προλάβαμε να κάνουμε όσα θα θέλαμε. δεν είχαμε περισσότερε μέρε. Πάντω ε, τη βρήκα πολύ διαφωτιστική την αποστολή αυτή και πρέπει να πω ότι μου άλλαξε και ε, αντίληψη για ορισμένα πράγματα. Με εντυπωσίασαν τα εξή λοιπόν. Πρώτον, απτό, απτό ήταν το ότι οι πολιτικοί συνομιλητές μας, οι υπεύθυνοι, ο Πρωθυπουργός, βουλευτές, φοβήθηκαν, φοβήθηκαν πάρα πολύ σε σχέση με το Ισλαμικό κράτος, όπως ε, θα μπορούσα να το πω μεταφορικά, πέρασε από δίπλα τους ένας Αρμαγεδόν. Έτσι λοιπόν έχοντας ε, υπόψη τις συνέπειες αυτών των επιθέσεων βλέπουμε και πώς ανταποκρίθηκαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν όλο και περισσότερο περιπέσει σε ε, διχασμούς είναι τώρα σε θέση να τους ξεπεράσουν, είναι να τους ξεπεράσουν γιατί είδαν την καταστροφή που θα σήμαινε το Ισλαμικό κράτος. Άρα βλέπουμε πολύ σημαντική ε, προσκόλληση σε αυτή την ιδέα του Ιράκ, της διαφύλασης ενός ε, κράτους ακέραιου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λόγω του φόβου αυτού του Ισλαμιστή που ήταν ο εχθρός του στο Ισλαμικό κράτος, αλλά ταυτόχρονα και με αλλαγή και της προσδοκίας και διεκδίκησης σε μια διακυβέρνηση, γιατί περί αυτού πρόκειται πλέον. Ζητούν να έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης του κράτους οι πολίτες και όχι μόνο ε, να είναι η διακυβέρνηση στα χέρια των Σιητών ή των Σουνετών ή των, ε, Τουρκμα, ε, Τουρκομάνων, αλλά να την έχουν οι πολίτες για το κράτος τους, εθνικό κράτος λοιπόν και όχι εσωτερική διχασμή. Ήταν το μήνυμα που μας απέστειλαν οι περισσότεροι ή όλοι οι συνομιλητές της επαφές μας και το βρήκα συναρπαστικό. Δεύτερο στοιχείο, το είπατε κι εσείς, εμείς οι Ευρωπαίοι στο Ιράκ μπορέσαμε να αναγνωρίσουμε ένα κράτος το οποίο θέλει και επιτρέπει την υπέρβαση στην ακραία πόλωση που γνωρίζουμε στην περιοχή μεταξύ Τουρκίας, Ιράν και Σαουδικής Αραβίας. Γιατί είναι θανάσιμη παγίδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση το γεγονός ότι καλείται να κάνει επιλογές εναλλάξ μεταξύ της μίας ή της άλλης χώρας. Σημαντικές και οι τρεις βεβαίως, καμία δεν πρέπει να αποκλειστεί, αλλά διαρκώς καλούμεθα να κάνουμε επιλογές εναλλάξ. Και σε αυτό έχουμε βρεθεί στο ίδιο μήκο κύματο με το Ιράκ, βεβαίω με άλλε προτιμήσει, ίσω με άλλη βαρύτητα σε κάθε περίπτωση, λόγω και τη γεωγραφική θέση, αλλά πάντω βλέπουμε ότι ξαναβρίσκει μια θέση το Ιράκ, όπως ε, την είχε άλλωστε και πριν από 15 χρόνια, την θέση μιας περιφερειακής δύναμης. Τελευταίο σημείο, και αυτό είναι το επίκεντρο των ανησυχιών που είχα πριν ε, φύγω για το ταξίδι. Είχα κάποιες αμφιβολίες πρέπει να πω, αλλά όταν ε, έχουμε μια τόσο έντονη επιρροή του Ιράν αφενός αφετέρου των Αμερικανών στο Ιράκ, η ανησυχία μου ήταν αν θα μπορούσαν οι Ευρωπαίοι να βρουν μια θέση και μετά το ταξίδι αυτό βλέπω από τις δύο πλευρές και από το Ιράκ και από την ευρωπαϊκή πλευρά ότι ναι, έχει θέση η Ευρώπη, έχει μια, ένα όραμα ευρωπαϊκό και για τα θέματα της ασφάλειας που μπορεί να προσφέρει και άρα μπορούμε να, να την ενισχύσουμε τη θέση αυτή. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ευκαιρία που προσέφερε αυτή η αποστολή. Δυσφορία μόνο η συντομία της μπόρεσε να προκαλέσει. Ίσως όμως έχουμε την ευκαιρία σε μια προσεχή ε, χρονική περίοδο, να δώσουμε και τη συνέχεια, να μην περιοριστούμε σε μία εφάπαξ επίσκεψη. Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί. Η διαδικασία είναι ευάλωτη. Θα μπορούσε ακόμα και να παρεκτραπεί γιατί μπορεί να επηρεαστεί από, οποιαδήποτε, από οποιουσδήποτε αστάθμητους ή ε, αντίξωους παράγοντες ανα πάσα στιγμή και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε και να την παρακολουθούμε. Ευχαριστώ Αγνώ, Γιάννα Γκόμες. Και εγώ αισθάνθηκα ιδιαίτερη ικανοποίηση από τα όσα είδαμε στο Ιράκ. Ε, ο Άγνο πολύ σωστά υπογράμμισε, ήταν πολύ σημαντική αυτή η μελέτη. Εγώ ήρθα στο Κοινοβούλιο το 4 σε μια εποχή όπου η περίοδο ήταν ε, διχασμένη μεταξύ Παλαιάς και Νέας Ευρώπης λόγω της ε, επίθεση στο Ιράκ και ανέλαβα το 2007-2008 την έκθεση για το Ιράκ, για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ. Και αυτή ήταν η πρώτη μου επίσκεψη στο Ιράκ. Μπόρεσα βέβαια όλα αυτά τα χρόνια να το ξαναεπισκεφθώ, όχι μόνο τη Βαγδάτη αλλά και άλλες ε, περιοχές και μπορώ να έχω μια εικόνα της εξέλιξης. Αυτό που μπορώ να πω ως κριτική για τις επισκέψεις αυτές είναι αφενός όταν πολυστομές και αφετέρου ότι τουλάχιστον δεν περιλάμβαναν τουλάχιστον το Ερμπίλ. Και επίσης ε, θα ήθελα να σημειώσω ότι βλέπουμε μία σύγκληση όλων των ε, εμπλεκομένων πλευρών, ύστερα από την αναγνώριση του κινδύνου στον οποίο εξετέθησαν τον κίνδυνο δηλαδή να αποτύχει το κράτος το ίδιο να καταληθεί και το την απειλή που αποτελούσε το Ισλαμικό κράτος που τους υποχρέωσε ως εκ τούτου να συγκλίνουν και να συνεργαστούν για την διάσωση της χώρας η οποία έχει βέβαια και κρίσιμο ρόλο για την περιφερειακή σταθερότητα και ισορροπία δυνάμεων όπως ε, συζητούσαμε νωρίτερα με τον ε, κύριο Πρέσβη κατηδίαν, ε, τον οποίο μάλιστα και ευχαριστώ για την εξαιρετική του δουλειά και την υποστήριξη που μας προσέφερε. Το Ιράκ λοιπόν, εάν κλείνει προς τη μία ή την άλλη πλευρά, δηλαδή εάν μπει στην περιφερειακή αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, θα μπορούσε να αποτελέσει και ρόλο αποσταθεροποίησης. Είναι πολύ σημαντικός, λοιπόν, πολύ πιο σημαντικός από ποτέ ο ρόλος του Ιράκ και νομίζω ότι μπορεί να μας ενθαρρύνει ε, η, ύπαρξη σημαντικών βελτιώσεων. Θα ήθελα βέβαια να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, άλλωστε μας το επεσήμαναν όλοι οι συνομιλητές μας, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων των μυστικών υπηρεσιών και της ασφάλειας, των υπηρεσιών ασφαλείας, αλλά και στη διαδικασία της εξομάλυνσης, στη δικαιοσύνη, που είναι απολύτω απαραίτητη για την εξασφάλιση ενός ορθώς λειτουργώντο ε, κράτου και, και βεβαίως και σε άλλα ζητήματα και για το πετρέλαιο και για την επίλυση των ε, κύριων ε, διαφορών για, τις, για τους φυσικούς πόρους, για το πετρέλαιο. Φερρυπίνει το ζήτημα του Κίρκουκ. Ε, μπορεί να διαδραματίσει λοιπόν ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ερώτησή μου προς τον πρέσβη Μπλεκουά είναι η εξή. Την πρώτη φορά που επισκέφτηκα εγώ το Ιράκ, Ε, με συγκλώνει στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν περιορισμένη στο βρετανικό συγκρότημα. Και ο πρόεδρος Σαλμαλίκη ε, μας είπε τώρα ότι υπάρχουν χώροι για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πρεσβεία που συγκεντρώνουν ε, εκπροσώπους χωρών που έχουν εντωμεταξύ αποχωρήσει, δεν έχουν πρεσβείες Βλέπω λοιπόν, να μην έχει αλλάξει τίποτα εντωμεταξύ, δηλαδή ούτε πολιτική βούληση φαίνεται να υπάρχει, ούτε πόροι κτλ. Αλλά τώρα και χωρίς να θέλω να επικρίνω τη χώρα. Βεβαίως και ήταν πολύ καλή και ευχαριστούμε ιδιαίτερως για τη φιλοξενία στο βρετανικό ε, συγκρότημα ή μπάνκερ. αλλά, αλλά μια και πρόκειται να αποχωρήσει με το Brexit κατά πάσα πιθανότητα το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επιδιώκει να έχει τις δικές της εγκαταστάσεις και εκεί να προσφέρει ε, στέγη και, σε και στα λοιπά κράτη-μέλη και στα κράτη-μέλη που δεν έχουν τα αυτόνομα, τις αυτόνομες εγκαταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιος ότι ο πρέσβης Πλεκού θα απαντήσει στην ερώτησή σου. Βεβαίω υπογράμμισες πως άπαξ και το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη χώρα θα, έχει, θα εμπέ, εμπίπτει και στην αρμοδιότητα της ΑΦΕΤ ως αρμόδιας καθήλυν επιτροπής για τις σχέσεις με τρίτες χώρες. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει να το επισημάνω ως πρόεδρος Επιτροπής, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι πρόεδροι άλλων επιτροπών που έχουν διαφορετικές απόψεις, όπως της Αλίας. Ο κύριος Μπούχνερ, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως ε, για πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να είμαι στην αντιπροσωπή αυτή. Ιδιαίτερος καλή αυτή η αποστολή. Ευχαριστώ θερμά λοιπόν. Πολύ καλή δουλειά. Πολύ δουλειά. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν και δεν θα τα επαναλάβω. Μια σύντομη παρατήρηση μόνο ότι με εντυπωσίασε η αισιοδοξία με όλες τις δυσκολίες που γνωρίζουμε και που βεβαίως τις συζητήσαμε διεξοδικά, με όλες τις δυσκολίες νομίζω ήταν σαφής ο, ε, η αισιοδοξία που εκφράσαν οι εκπρόσωποι του Ιράκ. Η οποία είναι και βάσιμη νομίζω. Διότι βλέπω ότι βελτιώνονται ιδιαίτερως οι οικονομικές προοπτικές της χώρας Πράγμα το οποίο κρίνω πολύ σημαντικό και που νομίζω ότι θα μπορούσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά τη να στηρίξει Φερρυπίν μέσω τη Επιτροπή Διεθνών, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τη ΣΥΝΤΑ. Έτσι λοιπόν ε, βλέπω εδώ μία προοπτική την οποία θα έπρεπε να υποστηρίξουμε περαιτέρω. Ο κύριος Μπούχνερ λοιπόν ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάρβερ τώρα. Ευχαριστώ πολύ ε, πήγα και πραγματικά χωρίς προκαταλήψεις και με εντυπωσίασε το πόσο ε, στρατευμένες είναι όλες οι πολιτικές ομάδες στο Ιρακινό Κοινοβούλιο υπέρ. Και νομίζω ότι από την τραγωδία αυτή, αν ε, έχουμε κάποια ε, θετικά θέματα, ε, είναι το γεγονός πως η τα πολιτικά κόμματα στο Ιράκ κατάλαβαν πως είχαν πολύ περισσότερα κοινά στοιχεία και συνεργάζονται πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν πριν από την εμφάνιση του ISIS και Κάτι το οποίο για μένα ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον, αναρωτικό και με έκανε να αισθάνομαι πιο σίγουρος είναι πως ε, γνωρίζουν πως έχουν πολιτιστικές διαφορές μεταξύ τους αλλά δεν θέλουν αυτό ε, να τους οδηγήσει σε περιφερειακές σειράξεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ελπιδοφόρο για το μέλλον του Ιράκ. Έχει πάρα πολλές ευκαιρίες και τώρα θα μιλήσω για το ΟΜΑΝ αλλά πριν περάσω εκεί Νομίζω ότι το Ιράκ θα μπορούσε να γίνει κάτι σαν το Ομάν στο μέλλον. Δηλαδή, ένα ουδέτερο σημείο σε μια περιοχή με αρκετή σταθερότητα. Αυτό είναι σημαντικό και θα ήθελα σε σχέση με το πώς είπε η Άννα να πω τα εξή. Βεβαίω η Αγγλία θα φύγει από, το, από ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό συμφωνούμε όλοι ανεξάρτητα με την ε, θέση μας. Έχει φτάσει μέχρι εκεί πια η κατάσταση. Όμως, ε, ξέρετε πως ε, μας πρόσκησαν πάρα πολύ από τη Βρετανική Πρεσβεία και εγώ θέλω να ξαναπάω και είναι μια ερώτηση που θέλω να σε απευθύνω και είχε ξαναγίνει ερώτηση αυτό από μερικά χρόνια. Είναι τι συμβαίνει και σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην πρωτοβουλία των 5i γιατί Ξέρετε πόσο ε, ανάγκη έχουμε αυτές τις ε, ξένες πρεσβείες. Και είμαι σίγουρος πως μετά τον Brexit η χώρα μου θα έχει πολύ καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ας φύγουμε από τις λεπτομερείς διευθετήσεις του τι ακριβώς πώς και τι θα τα οργανώσουμε. Νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα, η ασφάλεια, στα οποία, για τα οποία χώρη με ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Και νομίζω ότι στην επίσκεψή μας στο Ιράκ αυτό το είδαμε προφανέστατα και θα συνεχίσουμε ε, και εγώ θα συνεχίσω να στηρίζω όσο μπορώ ε, έτσι ώστε να μπορούμε να οργανώμαστε με το, τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζουμε τα κοινά μας ε, συμφέροντα σε τέτοιου είδους ε, περιοχές. Πάντως η Βρετανική πρεσβεία εκεί ήταν πάρα πολύ υποβοηθητική και νομίζω ότι Αντί να αγοράζει κτίριο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ιράκ, ας δώσει αυτά τα χρήματα σε κάτι άλλο που η χώρα το χρειάζεται περισσότερο. Αυτό. Και ας βασιστούμε σε αυτούς που κάνουν ε, αυτή τη δουλειά εδώ και χρόνια για να συνεχίσουμε να αισθανόμαστε αυτή την υποστήριξη. Σας ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις δεν έχουμε, οπότε νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω πάλι το λόγο για κάποια σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που όλοι σας, όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβαν το λόγο, κατανόησαν πολλά από τα εξαιρετικά περίπλοκα θέματα που έχει κατάσταση στο Ιράκ, τις προκλήσεις και νομίζω πως αν και η η επίσκεψη ήταν πάρα πολύ σύντομη. Ελπίζω πως δεν θα ήταν η τελευταία και θα μπορέσετε να ε, επεκτείνετε αυτή σας την εμπειρία. Πάντως τα πιο σημαντικά στοιχεία τα είδατε. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους σας να μεταφέρετε το μήνυμα αυτό, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Without the real experience, without being there, να πάει κανεί και δεν είναι εύκολο να αλλάξει κανεί την εικόνα που έχει το Ιράκ από τα προηγούμενα χρόνια και κυρίω από τι τραυματικέ εμπειρίε που προκάλεσε ε, ο Άισις για όλους μας, το Ισλαμικό κράτος, όχι μόνο για τους Ιρακινούς που ε, ένιωσαν άμεσα τις επιπτώσεις, αλλά και για τους Ευρωπαίους που έμαθαν να συμβιώνουν με την απειλή του Ισλαμικού κράτους στην καθημερινότητά τους. Και ξέρετε πως στο Ιράκ τελικά θα κερδιθεί η μάχη. Η κυρία Γκόμες έκανε κάποιες ερωτήσεις. όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σκοπό να αποκτήσει το δικό της κτηριακό συγκρότημα για την αντιπροσωπεία της στο Ιράκ. Αυτό ήταν πριν πάω εγώ αν θυμάμαι καλά, Όταν το Ισλαμικό κράτος είχε φτάσει στις πύλες Βαγδάτη ήταν πολύ δύσκολο να βρει κανείς εταιρείε που θα χτίσουν τέτοιου συγκροτήματα. Νομίζω πως η πρόταση βρίσκεται ακόμα στο τραπέζι. Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται το δικό της κτίριο, το δικό της χώρο, για το ρόλο που παίζουμε, για το πόσο ορατοί είμαστε. Έκτοτε, γιατί είμαστε στο Βρετανικό κόμπλεξ 9 χρόνια τώρα, αν δεν κάνω λάθος, η Βρετανική πρεσβεία μας έχει προσφέρει αυτό το ασφαλές καταφύγιο. Είναι μια πολύ καλά εξοπλισμένη βάση από την οποία μπορούμε εμείς να λειτουργήσουμε και όλοι. Ε, αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για τη στήριξη την οποία έχουμε λάβει μέχρι σήμερα και αυτό είναι κάτι που μας έχουν προσφέρει ε, ε, και έχουν προσφερθεί να το συνεχίσουν και μετά το Brexit για όσο χρειάζεται. Οπότε η απόφαση αυτή δεν είναι μια απόφαση που θα πάρω εγώ. Εγώ είμαι εκεί για να εφαρμόσω οποιασδήποτε οδηγίε λάβω και έχουμε ψάξει εναλλακτικέ λύσεις. Βέβαια θα πρέπει να δούμε τότε και τα οικονομικά θέματα. Είναι εξαιρετική χώρα ακριβά, ακριβή χώρα για να λειτουργήσει κανείς στο Ιράκ, λόγω ακριβώς των θεμάτων ασφαλείας που προκύπτουν. Και υπάρχουν και τα πρακτικά ζητήματα και τα επιχειρησιακά τα οποία θα πρέπει να στήσουμε. Επίσης μπορούμε να κάνουμε μία συνμίσθωση με κάποια άλλη χώρα. Δηλαδή αυτό μπορούμε να κάνουμε να μισθώσουμε κάποιες, κάποιους χώρους μαζί με τη γερμανική πρεσβεία. Είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει αλλά συγκεκριμένη απάντηση δεν έχω ακόμα. Πάντως η Βρετανική Πρεσβεία θα συνεχίσει να μας προσφέρει στήριξη και χαίρομαι που θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ε, προσφορά γιατί μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ ασφαλείς. Είδατε κι εσείς πώς γίνονται όλα. Και πραγματικά καταφέρουμε αυτή την περίπλοκη, το περίπλοκο καθήκον που έχουμε ε, αναλάβει να το φέρουμε σε πέρας, αλλά είναι ένας από τους στόχους μας για το μέλλον. Κύριε Μπούχνερ, για όσα είπατε περί οικονομίας, τελευταία παρατήρηση αυτή, είναι σίγουρα ένας από τους στόχους μας η ευημερία του Ιράκ ε, ε, ε, θα περάσει από την ανάπτυξη του ιδιωτικού κλάδου και από το γεγονός που θα πρέπει ο ιδιωτικός κλάδος να αποκτήσει ένα ρόλο στην ανασυγκρότηση με επενδύσεις, με περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. 60% του πληθυσμού είναι κάτω της ηλικία των, των 20 Οπότε ελπίζουμε πως με τη νέα αυτή συμφωνία ε, θα προσφέρουμε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπλέκουα. Ξέρω πως ο Υπουργό Εξωτερικών της Μαλαισίας έρχεται. Είναι στο διάδρομο, οπότε θα ήθελα να κλείσουμε με το Ιράκ και να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Λιωμαρή για το 27 να μας πει πώς πήγε η επίσκεψη στο Κατάρ και το Κουβέιτ. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και κάποια σχόλια για το Ομάν, αλλά νομίζω ότι γενικά μπορούμε να πούμε στο το Ομάν πήγε καταπληκτικά, εξαιρετική οικοδοσπότης, αισθανθήκαμε στο σπίτι μας για το 27. Ε, η συνάδελφος, ε, κύριε Πρέσβη, μπορείτε βεβαίως να μείνετε κοντά μας, αλλά ξέρω πως έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών. Ευχαριστώ πολύ, αφού μου το ζητήσατε προηγουμένως, θα πω δύο λόγια πολύ γρήγορα για το ΟΜΑΝ, γιατί θα έλεγα πως ε, νομίζω ότι εδώ μιλάμε για τους αντίποδες του Ιράκ. Δηλαδή χώρα, μία χώρα πολύ μικρή χώρα, μια χώρα η οποία έχει ελάχιστο ε, φυσικό πλούτο και είναι μια χώρα η οποία δεν έχει γνωρίσει τον πόλεμο. Είναι μια χώρα σχετικά σταθερή. Είναι μια χώρα η οποία ακολουθεί εσωτερική πολιτική, ε, εσωτερική πολιτική που βρίσκει μια ισορροπία μεταξύ της των παραδόσεων που βλέπουμε σε όλες τις ε, εκφράσεις της ζωής και ε, ενός σύγχρονου τρόπου ζωής που θα ακούσετε και στο τέλος της εβδομάδας, γιατί με κάλεσαν και μία συνδιάσκεψη ε, για το ΟΜΑΝ το 2040. Μιλήσαμε λοιπόν ε, για το ΟΜΑΝ και είπαμε ότι εκεί ε, ε, το Ισλάμ εκεί είναι αρκετά διαφορετικό. Υπάρχει ένας βαθμός θρησκευτικής ανοχής, αρκετά διαφορετική από τις όμορες χώρες και γίνεται αυτή τη στιγμή και μία προσπάθεια διαλόγου με το Ιράν. Το ΟΜΑΝ θα ήθελε να παίξει ένα διεθνή ρόλο, κυρίως στην δική του περιοχή, πιο ορατό. Προσπάθησε ή προσπαθεί να παρέμβει ε, στις διάφορες Ιράκες που υπάρχουν εκεί και στην Ιεμένη. Αλλά ξέρετε πως αυτό εκνευρίζει τη Σοδική Αραβία και εκεί βέβαια υπάρχουν πολλές τριβές. Είναι μια χώρα λοιπόν που αναπτύσσεται με σχετικά αρμονικό τρόπο ε, και σε εσωτερικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο και το μεγάλο ερωτηματικό είναι η αβεβαιότητα, η πολιτική αβεβαιότητα που έχει να κάνει με την διαδοχή του Σουλτάνου που έχει αρχίσει να είναι αρκετά ηλικιωμένο και δεν έχει ε, ορίσει επίσημα διάδοχο. Αυτά είχα να πω για το ΟΜΑΝ, δεν ξέρω αν αυτό ε, θέλατε και εσείς να ακούσετε, μια γενικότερη εντύπωση. Γρήγορα λοιπόν, θέλω να σας περιγράψω και το τι έκανε η αποστολή μας στο Κατάρ και στο Κουβέιτ, τέλη της περασμένης χρονιάς, γιατί νομίζω ότι συναντηθήκαμε και σε ένα αεροδρόμιο. Νομίζω εσείς επιστρέφατε από τη δική σας αποστολή στο Ιράκ. Και για το Κατάρ να πω το εξή. Οι σχέσεις μας με το Κατάρ είναι εξαιρετικές. Έτσι λοιπόν, σε ένα περιβάλλον φιλικό, ανοιχτό, αμοιβαίου σεβασμού, ε, κάναμε αυτή την επίσκεψη. του. πιο ενδιαφέρον ήταν να δούμε τις αλλαγές από τότε που πέρυσι, το 2017 δηλαδή, ε, κηρύχθηκε το εμπάργο από, κάποια, από κάποιες ε, χώρες των ε, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να σας πω πως αυτό το εμπάργο έχει να κάνει καταρχήν με το τι ε, θέλουν τα Εμμυράτα, τον Μπαχρέν και, το, ε, και η Σαουδική Αραβία, χώρες δηλαδή του κόλπου και πώς επηρέασε και ψυχολογικά και οικονομικά το Κατάρ. Η χώρα κατάφερε να ξεπεράσει τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν από το εμπάργο που κατάφερε να ξαναβρει ένα δυναμισμό στην οικονομία του και είναι τώρα πιο στεναρό οικονομικά, πιο ανοιχτό προς νέες χώρες με τις οποίες ανέπτυξε εμπορικές σχέσεις και όχι μόνο εμπορικές και κυρίως με το Ιράν, την Τουρκία και με κάποιες χώρες από την Ασία με τις οποίες έχει αυτή τη στιγμή ε, αναπτύξει στρατηγικές ε, σχέσεις, Τουρκία και Ιράν κυρίως, και τέλος βλέπουμε στο Κατάρ να έχει διατηρηθεί ο δυναμισμός της χώρας, να τρέχουν και κάποιες μεταρρυθμίσεις και να έχει ακόμα ένα διεθνή ρόλο. Μιλήσαμε πολύ για το εμπάργκο και για την κρίση στον κόλπο. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι προφανές πως μπορούμε να είμαστε κάποιο είδους αλλά δεν μπορούμε να αναλάβουμε διαμεσολαβητικό ρόλο. Μεταξύ του πρέπει να τα βρούμε, αλλά μπορούμε εμείς να είμαστε εγγυητή οποιασδήποτε λύση. Για να βοηθήσουμε στο μέγιστο να επιληθεί αυτή η σύραξη υπέρ της περιοχής εκεί, αλλά γιατί είναι και υπέρ των δικών μας συμφερόντων, υπέρ τη δικής μας σταθερότητα, ε, η οποία επηρεάζεται και από τη σταθερότητα στην περιοχή αυτή. Για τα μίντια να σας πω πως ε, κάλυψαν την επίσκεψή μας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κάναμε συναντήσεις με τη Σούρα, που είναι αν θέλετε ομόλογός μας, και μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τον πρόεδρο και μια αντιπροσωπεία ε, μελών αυτής, και μάλιστα μαζί τους, όπως και με τους υπόλοιπους συνομιλητές μας από την κυβέρνηση, μιλήσαμε πάρα πολύ για την κρίση αυτή και μας επανέλαβαν πως οικονομικά έχουν βγει από την κρίση, αλλά επέμεναν όλοι ε, στον αντίκτυπο που είχε το εμπάργο στην προσωπική ζωή όλων και το τι είχε να κάνει σε επίπεδο ιατρική περίθαλψης για παράδειγμα, τι είχε να, πώς επηρέασε του φοιτητέ και τι οικογένειε οι οποίε πολλέ φορέ ε, χωρίζονται από το εμπάργκο. Επίση, μετά συναντηθήκαμε με εκπροσώπους κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και όλοι ε, παρουσίασαν την ίδια περίπου κατάσταση και ασχολήθηκαν κυρίως με τις αρνητικές επιπτώσεις για τα μεμονωμένα άτομα, άτομα αυτού του εμπάργου. Και είπαν πως ικανοποιεί ιδιαίτερα η προσέγγιση, κυρίως η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο υπουργό Εργασίας ανακοίνωσε κάποιες αλλαγές για το μέλλον με αρκετές, αρκετούς νόμους που έχουν ως σκοπό να προστατεύσουν τους ε, αλλοδαπούς ε, εργαζόμενους όπως επίσης και για μια μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου. Και πιστεύω πως εδώ η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι πως αυτή η κρίση είχε το εξής αποτέλεσμα, να ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ το Κατάρ στην εικόνα που ε, έχει... Ε, που έχει και ε, σε αυτή την προσπάθεια του να έχει μια θετική εικόνα προσπαθεί να προσαρμοστεί σε κάποιους κανόνες και πρότυπα που ακολουθούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή που ακολουθούν άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Οπότε έχουν αναλάβει κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επόμενη λοιπόν συνάντηση τη διακοινοβουλευτική με το Κατάρ που θα γίνει μέσα το 2020 ε, είπαν ότι θα παρουσιάσουν κάποια μέτρα και επίσης μιλήσαμε για τη δυνατότητα Συγκεκριμένη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, Καταριανής Σούρα μεταξύ των διοικητικών μας υπηρεσιών και επιμένω εδώ είναι καλό και θα επιμείνω να υποδεχτούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν ε, αριθμό ε, υπαλλήλων της ε, Σούρα που θα ήθελα να δουν πώς εργαζόμαστε εμείς για να εμπνευστούν. Νομίζω πως θα πρέπει να αναλάβουμε και δράση για να συνεχιστεί ο διάλογος και ανταλλαγή ε, απόψεων με το Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Κατάρ και της ε, δικής μας, ε, των δικών μας επιτροπών και πιστεύω πως καλό θα ήταν να οργανώσουμε και συναντήσεις εδώ αυτά σε γενικές γραμμές για την επίσκεψη στο Κατάρ. Μάλιστα, μετά το Κατάρ πήγαμε στο Κουβέιτ. Ένα διήμερο περάσαμε και εκεί. Ε, και θα ήθελα να σας επισημάνω σημαντικό στιγμή, Εδώ και αρκετά χρόνια το Κουβέιτ ένιωθε κάπως εγκαταλελειμμένο, παραμελημένο. Και το γεγονός ότι έγινε ο διαμεσολαβητής στην κρίση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, το έκανε το Κουβέιτ να ανακτήσει την ε, αυτοπεποίθηση, την εμπιστοσύνη του και να παίξει ένα διεθνή ρόλο. Και γι' αυτό στηρίχθηκε στην αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να εμψυχώσουμε, να θαρρύνουμε το κουβέιτ, να διεκπαιρεώσει αυτό το θετικό του ρόλο είναι πολύ σημαντικό και το επιβεβαιώνει και σε σχέση με το περιβάλλον των γειτονικών χωρών. Είναι μεν μικρή χώρα το Κουβέιτ, αλλά ακριβώ έχει ικανότητα διαλόγου με τους πάντες. Και χάρη σε αυτή την ικανότητα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα το αναγνώρισε αυτό, γιατί όταν φτάναμε στο Κουβέιτ αποφασίσαμε να ανοίξουμε γραφείο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κουβέιτ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ε, τη στιγμή που το Κουβέιτ ε, δήλωσε ξεκάθαρα ότι η κάπως αλλοπρόσελη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών τους προβληματίζει και τους ανησυχεί ιδιαίτερα. Ως εκ τούτου, το Κουβέιτ θα ήθελε και μας έδωσε ως παράδειγμα την αποχώρηση των ε, Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Σύρια ε, θέλουν να αποστασιοποιηθούν κάπως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε αντιστάθμισμα θα ήθελα να πλησιάσουν πολύ περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι προφανές ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει εδώ σημαντικό ρόλο. Πολλό μάλλον, όπως σας είπα, που το ε, κοινοβούλιο του Κουβέιτ είναι το μόνο που εκλέγεται με άμεσες και δημοκρατικές εκλογές. Το μόνο κοινοβούλιο στην περιοχή που εκλέγεται με τέτοιο τρόπο, άμεσο και δημοκρατικό. Και αυτή η κατάσταση είναι πολύ ευνοϊκή για να αναπτύξουμε περισσότερες σχέσεις με τους ομολόγους μας στο Κουβέιτ. Ε, συναντήσαμε με πολλούς βουλευτές, μιλήσαμε για πολλά θέματα, όπως τα δικαιώματα των γυναικών, Ε, και το θέμα της εκλογής. Περισσότεροι εκλέγονται δημοκρατικά, πάντως υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Συζητήσαμε για τη θανατική ποινή, συζητήσαμε για το καθεστώς των απάτριδων, λεπιντούν όπως λένε εκεί, τους αλλοδαπούς ε, εργαζομένους ε, και ούτω καθεξής. Επίσης, μας υποδέχθηκε ο Εμμύρης, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, και όλοι υπογράμμισαν την επιθυμία τους να παίξουν ρόλο στη σταθεροποίηση της περιοχής. Επίσης, ε, εξέφρασαν την επιθυμία τους για στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί προτείναμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Η επόμενη διακοινοβουλευτική συνδιάσκεψη θα γίνει το 2020, αλλά προτείναμε και πιο συγκεκριμένη συνεργασία με διαπροσωπικές επαφές και συζητήσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, τη νέα νομοθεσία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα δύο ταξίδια, οι δύο αποστολές που είχαμε στο Κατάρ και το Κουβέ και στο Αμάν προηγουμένως. Ευχαριστούμε κυρία Λιωμαρή για την ενημέρωση που μας κάνατε για τις αποστολές αυτές. Ε, περιμένει πρώτο θεωρών ο Υπουργό Εξωτερικών της Μαλαισίας η κυρία Λόχπιλερ, ζήτησε το λόγο και μετά θα περάσουμε αμέσως στο επόμενο θέμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Εγώ θα μιλήσω για το Κατάρ, γιατί όταν ο Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ ε, ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μα εξήγησε τι μεταρρυθμίσει τις νομικές για τα δικαιώματα των, των μεταναστών. Επίσης μιλήσαμε ε, ε, για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ε, των μεταναστών και σε σχέση με τη FIFA. Πώς εφαρμόζονται όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι οι μεδαποί οι εργαζόμενοι ε, ξερούνται από αυτή τη νομική μεταρρύθμιση. Αλλά και στο Κατάρ εφαρμόζονται παρόμοιες ε, μεταρρυθμίσεις και γι' αυτό θα ήταν και αυτά τα θέματα ενδιαφέροντα για συζήτηση αργότερα. Αν το επιτρέπει φυσικά και ο χρόνος. Ευχαριστούμε. Άλλος κανείς δεν θέλει το λόγο. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το 28, και θα παρακαλέσω τον καλεσμένο μας, τον Υπουργό Εξωτερικών της Μαλαισίας, να καθίσει δίπλα μου. Right, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη τιμή θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό Εξωτερικών της Μαλαισίας, τον κύριο, και ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά του, τον κύριο Σαϊφουντίν Αμπτουλά. Εξοχότατε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχουμε μια τακτική συνεδρίαση, το πρωί είχαμε ψηφοφορίες και προχωρούμε στα υπόλοιπα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος ε, για την παρουσία εδώ και πριν σα δώσω το λόγο θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή. Ο υπουργό ε, στις 11 και 35 θα πρέπει να αποχωρήσει. Έχουμε μισή ώρα και κάτι. Ε, καταρχήν, μετά από μια έκθεση πρωτοβουλία του 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησε συστάσεις για τι διαπραγματεύσει Ευρωπαϊκή Ένωση Μαλαισία για μια συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία. Το Συμβούλιο πρότεινε ολοκλήρωση συμφωνία το 2018, αλλά τελικά τα συμβαλόμενα μέρη δεν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για το κείμενο. Ελπίζω τώρα να ε, υπογραφεί συμφωνία μέχρι το τέλη του έτους, δηλαδή έχουμε 11,5 μήνες για να το καταφέρουμε και να παραπευθεί το θέμα από το Συμβούλιο στο Κοινοβούλιο για να δοθεί η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακολουθήσαμε και τις εκλογές που έγιναν στη Μαλαισία το Μάιο, που για πρώτη φορά είχαμε επιστροφή της αντιπολίτευσης στο πολιτικό προσκήνιο και εντολή για σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Θα μας πείτε λοιπόν ποιο θα είναι το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης. Τι σχέδια έχει ο Πρωθυπουργό σα και ποιε είναι οι πολιτικές σας προτεραιότητες. Και μάλιστα πέρυσι είχαμε επισκεφθεί την περιοχή με μια αντιπροσωπεία πήγαμε στην Ινδονησία και την Ταϊλάνδη και επισκεφθήκαμε και την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος για την παρουσία σας και ελπίζω να περάσουμε, να έχετε ενδιαφέρουσες επισκέψεις στις Βρυξέλλες και επικοδομητικές συζητήσεις. Πάντως Ελπίζω να είναι και η Ευρώπη προτεραιότητα της κυβέρνησης στην Κουάλα Έχετε το λόγο. Σαλάμ αλέκουμ. Καλημέρα σε όλους σας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα που μιλώ σε αυτή την ομίγυρη. και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε από χθε έχω έρθει για τη συμμετοχή μου στην Υπουργική Διάσκεψη των χωρών ΑΣΕΑΝ. Είχαμε πολύ επικοδομητική συζήτηση καρποφόρα χθε το απόγευμα και συναντώ και ομολόγους μου, υπουργού Εξωτερικών ε, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλές διμερείς επαφές που θα έχουμε. Το Μάιο και πιο συγκεκριμένα στις 9 Μαΐου το 2018 για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια ανεξαρτησίας οι Μαλαισιανοί αποφάσισαν να αλλάξουν την ομοσπονδιακή τους κυβέρνηση. Τώρα έχουμε μια νέα κυβέρνηση τη οποία ηγείται μια νέα πολιτική συμμαχία, ένας νέος πολιτικός συνασπισμός, το Πακατάν Χαραπάν, στα αγγλικά θα το μεταφράζαμε ως «Η Συμμαχία της Ελπίδας», «Πακατάν Χαραπάν», «Η Συμμαχία της Ελπίδας». Ο Πρωθυπουργό σήμερα είναι ο Δόκτωρ Μαχαθήρ Μοχαμέντ. Θα τον θυμάστε πολύ. Ήταν και στο παρελθόν, διετέλεσε Πρωθυπουργό της Μαλαισίας για 22 χρόνια πριν αποχωρήσει από τον πολιτικό βίο για μία δεκαπενταετία, άφησε το παλιό του κόμμα, σχημάτισε, ίδρυσε ένα νέο κόμμα και σε συνεργασία με άλλα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης δημιούργησε ένα συνασπισμό. Για παράδειγμα το κόμμα της δικαιοσύνης του Ανώ Ιμπραχήμ. Μερικοί α, ε, μπορεί να το γνωρίζετε, το θεωρείτε παλιό φίλο. Το κόμμα της δημοκρατικής δράσης επίσης του Λίγκου Ανέγκ που είναι τώρα υπουργό Οικονομικών. Ενώ ο Ανώ Μπραχήμ θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργό. Τουλάχιστον αυτό προβλέπει η συμφωνία ε, του σχηματισμού της νέας κυβέρνησης ε, που απαρτίζεται από κόμματα του συνασπισμού. Και το τέταρτο κόμμα είναι το Αμάνα, ένα μουσουλμανικό φιλελεύθερο κόμμα. Είναι το κόμμα των μουσουλμάνων δημοκρατών. Είναι προοδευτικό κόμμα, μουσουλμανικό, με προοδευτικό δε, ανοιχτό όμως και προς μη μουσουλμάνους. Είναι κάπως διαφορετικό μουσουλμανικό κόμμα, πιο ανοιχτό. Και μάλιστα το βασικό μα σύνθημα στην προεκλογική εκστρατεία ήταν η πάταξη της διαφθοράς. Και την ώρα που σας μιλώ, ο Πρωθυπουργό Μαχατήρ ε, βρίσκεται στη Βιέννη και ομιλεί σε μια διεθνή διάσκεψη για την πάταξη της διαφθοράς. Επίσης, ε, προτείναμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα πολλές μεταρρυθμίσεις και μερικές από αυτές προσπαθούμε να τις δρομολογήσουμε. Για παράδειγμα, τη μεταρρύθμιση ε, για, και συνιστούμε πολλές επιτροπές για την ε, χάραξη πολιτικών και ορίζουμε ε, δικαστές, διορίζουμε δικαστές επικεφαλής των αστυνομικών σωμάτων. Αυτή είναι μια πολιτική μεταρρύθμιση. Άλλη μεταρρύθμιση θα είναι εκλογική μεταρρύθμιση. Ε, ορίσαμε νέο τρόπο της ε, εκλογικής, νέο πρόεδρο της εκλογική επιτροπής. Έχουμε κάποια προβλήματα με την συνταγματική αναθεώρηση, γιατί δεν εύκολα να συγκεντρώσουμε την πλειοψηφία που απαιτείται γι' αυτό. Κάνουμε πάντως ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε τουλάχιστον δύο βασικά θέματα του παρελθόντος. Ε, δύο ζητήματα που δυσκολεύουν τις εκλογές. Ε, και κυρίω στην σημερινή κυβέρνηση. Θέλουμε λοιπόν να πραγματοποιήσουμε αυτές τις ε, νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, ε, θεσπίσαμε δικαιοστάσιο μορατόριο για τη θανατική ποινή. και θα καταργήσουμε και το νόμο για τη θανατική ποινή, το νόμο που ε, περιορίζει την ελευθερία του τύπου, την πολυφωνία και θα μεταρρυθμίσουμε πολλές νομοθεσίες ε, ενώ θα καταθέσουμε και νέα νομοθετήματα. Έχουμε το νέο νόμο της αρμονίας που λέμε, που ουσιαστικά καταπολεμά τις διακρίσεις. Θέλουμε όλες οι πολιτικές μας να είναι συμμετοχικές, ε, να μην αποκλείουν κανέναν Μαλαισιανό. Γιατί η Μαλαισία ε, έχει πολλές, απαρτίζεται από πολλές φυλές, εθνότητες και θρησκείες και θέλουμε αυτή την πολυμορφία να τη διαφυλάξουμε. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μια απόπειρα να σταματήσει η ρατσιστική πολιτική, γιατί ο ρατσισμός δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ οξύ στη Μαλαισία, αλλά υπάρχει πρόβλημα ρατσισμού. Και υπάρχει πρόβλημα γιατί ο ρατσισμός και οι πολιτικοί έχουν τόσο βαθιές ρίζες ε, και είναι τόσο ε, στην κοινωνία που μερικοί δεν το αντιμετωπίζουν ως πρόβλημα. Και αν πει κανείς θέλει να ξεριζώσει την ρατσιστική πολιτική, μερικές φορές αντιμετωπίζουν τον ίδιο ως πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα και να δημιουργήσουμε κίνητρα για τους πολιτικούς ε, ε, να καταπολεμήσουν το ρατσισμό και να μην επικεντρώνονται σε μία φυλή μόνο ή σε μία θρησκεία μόνο. Θέλουμε να έχουμε μία ευρύτερη προοπτική και όχι μόνο θρησκευτική ή μόνο ρατσιστική. Επίσης, ε, πασχίζουμε για να ξαναβάλουμε σε θετική πορεία την οικονομία μας. Πριν τις τελευταίες εκλογές είχαμε βαρύτατο χρέος, μεγάλο χρέος πάνω από 800 δισεκατομμύρια. Όταν αναλάβαμε όμως ε, τα καθήκοντά μας και κοιτάξαμε τα λογιστικά ε, βιβλία, είδαμε ότι το χρέος δεν ήταν 800 δις, αλλά 1,3 εκατομμύρια, που είναι τεράστιο ποσό για μια μικρή χώρα σαν τη Μαλαισία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε νέες ρυθμίσεις. Ε, θα πρέπει να αναδιαπραγματευτούμε κάποιες συμβάσεις που έχουμε με αλλοδαπές ε, εταιρείε, κυρίως κινέζικες. Και προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τώρα κάποιες συζητήσεις και τέτοιες ρυθμίσεις. Η νέα κυβέρνηση έχει αναλάβει δέσμευση και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ήδη διορθώσει. Είχε μάλλον ήδη κυρώσει τρεις από τις εννέα βασικές ε, διεθνείς συμβάσεις για τα παιδιά, για τις γυναίκες και για τα άτομα με αναπηρίες. Έξι ακόμη διεθνείς συμβάσεις θα πρέπει να κυρώσουμε προτεραιότητά μας είναι να κυρώσουμε τη σύμβαση κατά των βασανιστήριων και των αναγκαστικών εξαφανίσεων. Και θα είναι δύσκολη αυτή η διαδικασία, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τη διεκπαιρεώσουμε. Και θα δούμε πώς θα υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Μακάρι να μπορούσα να σας ε, ανακοινώσω την κύρωση και άλλη σημαντική διεθνούς σύμβασης, αλλά για λόγους τακτικής δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει πρώτα να γίνει στέψη του νέου βασιλέως. Θα φαντάζεστε για ποια σύμβαση σας μιλώ, για ποια διεθνή συνθήκη. Σας άφησα κάποια υπονοούμενα. Στι 31 Ιανουαρίου θα λάβει χώρα η στέψη του νέου βασιλέω. και τότε θα κάνουμε και την ανακοίνωση. Και τότε ίσως μπορέσουμε να μοιραστούμε μαζί σας τις ε, νέες αποφάσεις. Πάντως είμαστε προσιλωμένοι στην τήρηση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδουμε στις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Μαλαισίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δεσμοί μας είναι ιδιαίτερα ισχυροί στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Επίσης, οι δύο πλευρές έχουμε ουσιαστικές και βαθιές διμερείς σχέσεις στις ε, αξίες των ανθρωπινών δικαιωμάτων, αλλά και σε μια σειρά από διεθνή ζητήματα συμφωνούμε. Έχουμε επισκέψεις ψηλού επίπεδου μεταξύ Μαλαισίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταλλαγές επισκέψεων, όπως επεσήμανε και ο Πρόεδρος. Και η ενίσχυση των σχέσεων αντικατοπτρίζει οπωσδήποτε τις αμοιβαίες σχέσεις, αλλά και τον, ε, την παγκόσμια αντανάκλαση μας, ε, τον απόϊχο αυτών. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία ως διεθνής ε, εμπορικός εταίρος η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Μαλαισία τελευταία πενταετία. Θέλουμε να καλέσουμε περισσότερους Ευρωπαίους επενδυτές για την ε, διερεύνηση νέων δυνατοτήτων, για τη γεωργία, την αυτοματοποιημένη τεχνολογία, την ε, ε, πληροφορική και άλλα ζητήματα στη Μαλαισία. Κάποιες συμφωνίες ήδη διαγράφονται και εμείς από πλευράς μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κλείσουν κάποιες από τις λεπτομέρειες των συμφωνιών ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς ε, τους αξιότιμους κυρίες και κυρίους ε, βουλευτές του σώματος για το θέμα του φινικελαίου. Ερχόμενοι στις Βρυξέλλες ε, φέραμε μαζί μας την πεποίθηση πω θέλουμε να ενισχύσουμε τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και ΑΣΕΑΝ ως κράτος μέλος ΑΣΕΑΝ, αλλά και ως ΑΣΕΑΝ συνολικά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε να αναβαθμίσουμε το ρόλο μας ως απλώς, ε, από απλώς εταίρου διαλόγου σε στρατηγικού εταίρου. Αυτό είναι στόχος μας. Ταυτόχρονα όμως, ε, και αυτό το υποστηρίζουν και τα άλλα κράτη του ΑΣΕΑΝ, η Μαλαισία θέλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει αυτό το ζήτημα του φινικελαίου ως σημαντικό. Είχαμε κάποιες συζητήσεις. Δεν μπορώ να πω ότι έγινε πραγματικός διάλογος, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα να αντιληφθεί κανείς ποιες είναι οι θέσεις μας. Βεβαίως και εμείς σεβόμαστε τις θέσεις των άλλων Εχθές πρέπει να σας πω ότι δεν έγινε τίποτε το θεαματικό. Ε, πυροτεχνήματα δεν είδαμε και σε αυτό δεν φταίει ο χιονιάς. Αλλά σας διαβεβαιώ πως και η ΑΣΕΑΝ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, προσιλωμένες στην αναβάθμιση του καθεστώτος. Αποφασίστηκε χθε λοιπόν να αναβληθεί αυτή η αναβάθμιση. Θα εργαστούμε σκληρά από πλευρά ΑΣΕΑΝ αλλά και ιδιαίτερω η Μαλαισία και η Ινδονησία. Καλωσορίζουμε την ε, θέσπιση μια ειδική επιτροπή ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΣΕΑΝ για την εξέταση των ζητημάτων των σχετικών με το φινικέλαιο, έτσι ώστε να επιληθούν τα ζητήματα και να βελτιωθεί το χειρότερο δυνατό η κατάσταση. Αυτό βεβαίως είμαι στη διάθεση για να απαντήσω στις ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Και όπως είπαμε, είμαστε νέα κυβέρνηση, 8 μήνες μόλις, έχουμε αναλάβει καθήκοντα και κάνουμε σκληρή δουλειά για να βελτιώσουμε την κατάσταση περιλαμβανομένων των σχέσεων βέβαια Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαλαισίας αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασίας γενικότερα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε να συνεχίσουμε και κάποιες από τις οικονομικές μας, ε, από τις προσπάθειες για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ, εξοχότατε, για την ε, ομιλία, για την ε, παρουσίαση της κατάστασης στη Μαλαισία. Κάποιοι συνάδελφοι ασφαλώς θέλουν να λάβουν το λόγο. Πριν όμως δώσω το λόγο στους πρώτους που έχουν στήσει το λόγο, ο κύριος Λάγκεν, πρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας που είναι αρμόδια για τις σχέσεις με, την, ε, με τις χώρες της Ασίας. Είναι εδώ παρόν λοιπόν. Και ακούμε πρώτα τον κύριο Καν. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, Υπουργέ των Εξωτερικών, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι ιδιαίτερως για την παρουσία εδώ. Να, πω κάποιοι ξαναγυρνούν στην πολιτική. Γι' αυτό για κάποιους από εδώ μέσα που ίσως θα ήθελαν να, ή σκέφτονται να βγουν στη σύνταξη. Ίσως έχουν κάποια ελπίδα να ξαναγυρίσουν στο πολιτικό πεδίο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω για τους νόμους περί των στάσεων και πολύ σωστά είπατε με ικανοποιεί ιδιαίτερο ότι μιλήσατε για ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, αλλά δεν μιλήσατε για την ε, κατάργηση, εν πάση ουσιαστική αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικής με, την, με το έγκλημα τη τάση. Επίσης το ΑΖΕΑΝ. Είστε μία από τις 10 ε, χώρε ίσως και η μόνη που μίλησε ξεκάθαρα για την κατάσταση που αντιμετώπισε η κοινότητα των Οιγούρων στην ε, Κίνα, ε, ενώ το ΑΣΕ, η ΑΣΕΑΝ οργάνωση είχε μια πολύ επιφυλακτική στάση για την περιοχή των Ροχίνγκα στην ε, Μιανμάρ και τους εκτοπιστέντες. έχει υποδεχθεί πάρα πολλού. Γιατί λοιπόν και εσεί ω χώρα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Το Μαγκλαντές έχει υποδεχθεί πάρα πολλου Ε, γιατί λοιπόν και εσει ως χώρα γειτονική δεν δέχεστε περισσότερους, δεν προσφέρετε περισσότερη βοήθεια. Η κατάσταση εκεί πέρα είναι ε, καταστροφική, κατάσταση στο Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λόχπιλαρ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ τον Υπουργό Εξωτερικών ε, μίλησε ξεκάθαρα και έχει προβεί σε πρωτοβουλίες για την αλλαγή της κατάστασης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Χαίρομαι που ακούω πως καταργείται η θανατική ποινή. Τον επόμενο μήνα άλλωστε θα γίνει εδώ στις Βρυξέλλες το Παγκόσμιο Συνέδριο για την Κατάργηση Θανατικής Ποινής και με χαρά θα δούμε να λαμβάνει και η δική σας χώρα την πρωτοκαθεδρία στον αγώνα αυτό. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω σε πολυμερείς τομείς ή χώρους συναντήσεως όπως τα Ηνωμένα Έθνη, χώρους συνομιλιών, φόρα δηλαδή διεθνή, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, τι σκοπεύετε να πράξετε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σκοπευεται να πραξετε η ευρωπαικη ενωση παραδειγματι στη Γενική Συνέλευση, κατέθεσε μια πρόταση για ένα δίκτυο κρατών που θα μπορούσαν να μιλούν ε, με καλές επιδόσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα προέβαλαν ζητήματα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου θα είχε ιδιαίτερη σημασία να ε, ενσκύψουν τα Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστώ πολύ, Αναγκόμες. Στείλε τα τα παπά και ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Εξαιρετικές οι αλλαγές, απίστευτες οι αλλαγέ που βλέπουμε να παρουσιάζονται στη χώρα σας, ιδιαίτερα ε, το δικαιοστάθισιο στη θανατική ποινή που παρουσιάσατε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για το φινικέλο που ξέρω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη Μαλαισία, την Ινδονησία και τις λοιπές χώρες σας, εάν ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι θεσπίστηκε αυτή η ομάδα μεταξύ ε, των κρατών ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΑΣΕΑΝ ε, στο πλαίσιο των Εθνών. Πιστεύω ότι θα, μας επιτρέψει, θα σας επιτρέψει καταρχάς εσάς να ξεπεράσετε την εξάρτηση από την παραγωγή αυτή και σε όρους βέβαια απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα ξέρετε ότι εδώ στην Ευρώπη ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία ως προς τις ε, συνέπειες για το περιβάλλον της ε, παραγωγής φινικελαίου, αλλά και άλλα ζητήματα. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει κάποια πρόοδος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το όρομα, όραμά σα για την Κίνα πέραν των ζητημάτων των σχετικών με του Ουιγούρου που έθεσε και ο κύριο Κάνος, συνάδελφο. Οι προκλήσεις ε, που συνεπάγεται η στάση αυτή της επιβράδυνση τη που ονομάζεται Κίνα ε, στην περιοχή αλλά και ευρύτερα και όχι μόνο λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας της από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή αλλά και για, λόγω της έντονης παρουσίας της στις ε, νότιες σχετικές θάλασσες επίσης τους Ροχίνγκα. Τι έχετε να μας πείτε για τη σύγκρουση εκεί Η κυβέρνησή σας, από ό,τι μαθαίνω, σκοπεύει να ε, καταπολεμήσει τη διαφθορά. Να, υπήρχε ένα μεγάλο σκάνδαλο για την Goldman Sachs Είναι λοιπόν απαραίτητο να το παρακολουθήσουμε αυτό. Εμείς οι Ευρωπαίοι θα είμαστε διατεθειμένοι και να σας υποστηρίξουμε αλλά και να διδαχθούμε από την εμπειρία σας. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ και εν τέλει παρακαλώ τον Πρόεδρο της ε, Αντιπροσωπείας ΑΖΕΑΝ, κύριο Λάγκεν, να λάβει το λόγο. Πρόεδρε ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να έρθω εδώ ως ε, φιλοξενούμενος στην Επιτροπή σας και να λάβω το λόγο. Ευχαριστώ τον Υπουργό των Εξωτερικών και για την εκπροσώπηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αναλάβει εκ μέρους της ΑΣΕΑΝ γιατί έχει τώρα την Προεδρία η Μαλαισία. Η Μαλαισία λοιπόν ε, εκπροσωπεί ολόκληρη την περιοχή ΑΣΕΑΝ είναι μια χώρα η οποία μπορεί χάρη σε αυτή τη δημοκρατική επανάσταση και την στροφή προς τη δημοκρατία να αποτελέσει υπόδειγμα. Το δεύτερο διάγραμμα που μας παρουσιάζεται, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι υλοποιεί όλες τις προσδοκίες και υποσχέσεις που περιμέναμε και εμείς και ο λαός σας και όλοι ε, γύρω από τη Μαλαισία να δουν ε, τους τελευταίους 8 μήνες βλέπω να υλοποιείται ένα, ιδε, ένα ιδεώδες, ένα ορόσημο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την κοινοβουλευτική δημοκρατία και για τη δικαιοσύνη, η κατάργηση της ανατικής ποινή. Όλα αυτά βλέπουμε να είναι πράγματα στα οποία προσβλέπουν πάρα πολλές χώρες της ασιατικής περιοχής και των οποίων υπολείπονται πολύ. Και σε αυτό θέλω να τονίσω ιδιαίτερο, γιατί βλέπουμε με λύπη μα ότι υπάρχουν άλλε χώρε οι οποίε μάλλον οπισθοδρομούν. Γιατί στην Ταϊλάνδη, παραδείγματι, μπορεί να γίνονται εκλογέ και υπάρχει ένα σύνταγμα, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί κανεί να θεωρήσει και αμφισβητήσιμο. Αλλά στην Καμπότση απαγορεύονται οι εκλογέ. 45% ε, των ε, ε, αξιωμάτων αναγκάζονται σε παρέτηση των αξιωματούχων, αναγκάζονται σε παρέτηση λόγω αυτή τη. Ε, βγαίνουν εκτό αξιώματο λόγω αυτή τη τροποποίηση του συντάγματο. Και αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ λυπηρό και ενισχυτικό. Τώρα για το Φινικέλο, θα γνωρίζετε ασφαλώ ότι η αντιπροσωπεία ΖΕΑΝ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στο πλευρό σα 100%, στο πλευρό το δικό σα και τη Ινδονησία. Δεν αντιλαμβανόμαστε κάποιε κινήσει που έχουμε παρακολουθήσει και είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε στην ε, αντικειμενική και επιστημονική αξιολόγηση του φινικελαίου και με την αύξηση των ποσοτήτων των ποσοστώσεων εισαγωγής ε, με βάση και την οδηγία για την ε, ενέργεια. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, το έχουμε άλλωστε συζητήσει και διμερώς ε, το 95% της παραγωγής φινικελαίου προέρχεται από τι δύο αυτέ χώρε. Πώ μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να αναπτυχθούν διεθνεί προδιαγραφέ, πρότυπα δηλαδή, γιατί έτσι μπορούν να δοθούν και απαντήσει αποφασιστικέ σε πολλά από τα ερωτηματικά που έχουν διατυπωθεί για την παραγωγή του φινικελαίου. Είναι κάτι που συζητήσαμε και στην προηγούμενη σα επίσκεψη και θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει κάτι περισσότερο. Και μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με τις ε, τη νότια κινέζικη θάλασσα. Ε, φαίνεται πως υπάρχει μια ηρεμία παρότι το Βιετνάμ έχει κάποιες διαφορές ακόμη με την Κίνα, το Νότιο Βιετνάμ, το Βιετνάμ. Ε, το ζήτημα της οικονομικής συνεργασίας ε, στην περιοχή ΑΖΕΑΝ, πώς το βλέπετε, θεωρείτε δηλαδή ότι προχωρεί ένα επιτυχημένο εγχείρημα μέσα σε ένα σύντομο διάστημα, 5-10 χρόνια μπορούμε να δούμε την ε, επιτυχία του εγχειρήματο αυτού ή θα χρειαστεί να περιμένουμε περισσότερο. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ και βεβαίως προσβλέπουμε σε πολύ καλές σχέσεις Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λάγκεν. Ο υπουργό. Σας έχουν διατυπωθεί πολλές ερωτήσεις, πολλά ακόμα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, αλλά μια και δεν έχετε πολύ χρόνο ακόμη, σας δίνω το μικρόφωνο και παρακαλώ να μας πείτε δύο λόγια για το Ιναζεάν και τη... τι θα έλεγε η Μαλαισία σε περίπτωση που θα ήθελε να ενταχθεί το Ανατολικό Τιμόρ. Μια και έχουμε και προσκεκλημένο τον πρόεδρο. Είχαμε τον πρόεδρο του Ανατολικού Τιμόρ εδώ πριν από μερικούς μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω λοιπόν με τη δική σας ερώτηση, μια και είναι και πάρα πολύ σημαντική και έχουμε ξεκάθαρη θέση. Είμαστε υπέρ του Τιμόρ Λέστε ως μέλος της ΑΣΕΑΝ. Και μιλάμε με τα υπόλοιπα μέλη έτσι ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εξοχότητες για όλες τις ε, ερωτήσεις που μου απευθύνατε και θα προσπαθήσω να απαντήσω τις περισσότερες, αν όχι όλες. Έχουμε ένα-δύο μιλητές οι οποίοι έθεσαν θέματα τα οποία ε, αφορούν τους υπόλοιπους. Για την νομοθεσία Έχουμε επιβάλει ε, ένα ε, μορατόριο και την νομοθεσία με τις, ε, σχετική με τις στάσεις ο Γενικός Εισαγγελέας τον περασμένο μήνα, παρόλο που υπήρχε μια υπόθεση η οποία ε, μάλλον η δίωξη πρόκειται να ασκηθεί υπό αυτές τις κατηγορίες, αποφάσισε να μην χρησιμοποιηθεί ε, αυτή παρά να χρησιμοποιηθεί ο, ε, ο κώδικας ποινικού δικαίου. Γιατί εκτός ότι είναι απαρχιωμένη η σχετική νομοθεσία, είναι και πάρα πολύ αυστηρή και υπάρχουν και άλλοι νόμοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που χρειάζεται να απαγγελθούν ε, κατηγορίες. Οπότε ναι, έχουμε ξαναξεκινήσει τις προσπάθειες και η, πράξη, η νομοθετική πράξη περιστάσεων ε, είναι μία από αυτές τις οποίες προσπαθούμε να καταργήσουμε και ελπίζουμε θα καταφέρουμε ε, στην ε, επόμενη συνεδρίαση ε, που ξεκινά το Μάρτιο. Για τους Ροχίνγκα το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Κοιτάμε την κατάσταση και προσπαθούμε να κινηθούμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η θέση μας να είναι πιο σαφής και αν χρειαστεί να λάβουμε κάποιες αποφάσεις, να το κάνουμε. Για τους Ροχίνγκα, έχουμε τρία βασικά ζητήματα. Καταρχήν, εμείς συντασσόμαστε με την ε, διεθνή κοινότητα και ζητούμε οι αυτοργοί να δικαστούν. Εδώ έχουμε προσθέσει κάτι ακόμα και αυτό έχει να κάνει με την υπηκότητα. Δηλαδή, θα πρέπει αυτό να λαμβάνεται υπόψη ως μεγάλος και σημαντικός ε, παράγοντας τη στιγμή της ε, διαδικασίας συμφιλίωσης για μια βιώσιμη ειρήνη. Επαναπατρισμός. 700 με 800 χιλιάδες ροχίνγκα είναι στον Μπαγκλαντές και εκατοντάδες χιλιάδες στην ίδια τη Μαλαισία. Και πρέπει να σου πω πως έχουμε ανοίξει εμείς, για παράδειγμα, ένα νοσοκομείο στο Μαγκλαντές για τους ανθρώπους αυτούς. Πολλές χώρες του ΑΖΕΑΝ το κάνουν ε, με τον ίδιο τρόπο. Ε, και επαναλαμβάνω ότι έχουμε και αντίστοιχα ε, νοσοκομεία ε, και στα στρατόπεδα που συγκεντρώνονται οι άνθρωποι αυτοί στη Μαλαισία. Ε, προσπαθούμε να δούμε το θέμα της σχολικής εκπαίδευσης και βέβαια το πιο δύσκολο είναι να βγάλουν άδεια Για όσους πρόκειται να επαναπατριστούν από την Ταϊλάνδη, Νομίζω ότι θέλουμε να πείσουμε τη Μιανμάρ να μας επιτρέψει να κάνουμε περισσότερο. Αυτό θα είναι σε θελοντική ε, βάση, πάντα οι επαναπατρισμοί, με αξιοπρέπεια ε, και με βέβαια επεφρασμένη βούληση. Δηλαδή θα πρέπει να ζητήσουν οι Ροχίνγκα να επαναπατριστούν οι ίδιοι. Και εκεί ε, υπάρχει το έλλειμμα εμπιστοσύνη γιατί φοβούνται τι θα του συμβεί, δεν ξέρουν ποιο θα είναι το μέλλον του. Οπότε αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών ΑΖΕΑΝ είναι να βοηθήσουν βοηθήσουν την Μιανμάρ με την όλη διαδικασία επαναπατρισμού. Πρέπει να σας πω πως το πιο δύσκολο θέμα αυτή τη στιγμή με τους ε, πρόσφυγες που είναι ροχίνγκα είναι ότι δεν εμπιστεύονται τη χώρα τους και είναι πολύ δύσκολο να τους πείσει κανείς πως πλέον είναι ασφαλείς και μπορούν να επιστρέψουν. Το τρίτο θέμα είναι η ανθρωπιστική διάσταση στην οποία και αυτή αναφέρθηκα και εκεί προσπαθούν τα κράτη-μέλη της ΑΣΕΑΝ αλλά και η ΑΣΕΑΝ μαζί να λύσει ε, κάποια προβλήματα, να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για το θέμα ε, στο οποίο αναφερθήκατε που είναι η διάσκεψη για τη θανατική ποινή που θα γίνει στις Βρυξέλλες. Ο Υπουργός κ. Βικέλιου θα έρθει και μάλλον θα λάβει το λόγο και κατά τη διάρκεια της ε, διάσκεψης αυτής. Για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΖΕΑΝ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Μαλαισία και οι συζητήσεις που γίνονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήρθα σε... είχα συναντήσεις με κάποιους από τους επιτρόπους δύο από τους αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως έχω πει και στο παρελθόν και θα το επαναλάβω τώρα έχουμε αναλάβει τη δέσμευση και νομίζω ότι για πάρα πολλά θέματα ε, συμφωνούμε. Πολλά μπορούμε να κάνουμε για να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θρησκευτική ελευθερία. It is one of the that some of uh, Είναι κάποια από τα θέματα ε, τα οποία αυτή τη στιγμή συζητάμε ε, σε επίπεδο ΑΖΕΑΝ και για τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δική μου σύσταση είναι ένα από τα σημεία τα κομβικά για τις επιτροπές και τους επιτρόπους που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι να η σχέση τους με την Επιτροπή, τη Διακυβερνητική Επιτροπή της ΑΣΕΑΝ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και βεβαίως μπορούμε να μιλήσουμε και με την, ε, την κοινοβουλευτική διάσκεψη της ΑΣΕΑΝ και να σας φέρω εγώ σε επαφή με κάποιους από τους βουλευτές εκεί. Ήδη εκεί Ήδη εκεί συζητάνε κάποια θέματα ε, με το IPP ε, Οπότε κάνουν κάτι αντίστοιχο με εσά. Και για το φινικέλαιο να σας πω πως είναι μια μακριά ιστορία, το είδαμε και με τις είπα. Λοιπόν, είναι η μάχη μεταξύ φινικελαίου ε, και σόγιας. Και νομίζουμε πως κερδίσαμε, αλλά τώρα η κατάσταση είναι ακόμα πιο περίπλοκο, οι τάσεις όμως είναι παρόμοιες. Δηλαδή έχουμε τους, τα λόμπι, τα μίντια, κάποιους πολιτικούς και το καταλαβαίνω. Είμαστε πολιτικοί κι εμείς και ξέρουμε ε, σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες ε, τα λόμπι είναι πολύ ισχυρά και μιλάνε μια πολύ ισχυρή γλώσσα. Γνωρίζουμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να προσπαθήσω όμως πολύ σύντομα να σας πω το εξής. Για κάποια ζητήματα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Για παράδειγμα, αποψήλωση. Αυτά ε, είναι θέματα τα οποία έχουμε λάβει ε, πάρα πολύ ε, υπόψη και δεν πρόκειται να αποψηλωθούν άλλα δάση για να γίνουν καλλιέργειες. Ε, μπορούμε βέβαια να δούμε τι θα γίνει με την βιώσιμη παραγωγή, με την αύξηση παραγωγής σε ήδη φυστάμενες γέες έτσι ώστε να έχουμε την πιστοποίηση, για παράδειγμα, το ότι το φινικέλο που παράγουμε είναι βιώσιμο, είναι μια μαλαισιανή πιστοποίηση η οποία ε, θα ακολουθεί τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα. Έχουμε ήδη δεσμευθεί υπέρ των στόχων ε, βιωσιμότητας ε, για το 2030 και το έχουμε ήδη στο δικό μας αναπτυξιακό πρόγραμμα ε, για την περίοδο 2016-2020, το οποίο διανύουμε τη δεύτερη περίοδο και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς. Βέβαια, το θέμα είναι το εξή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάπου απαγόρευση. Όταν όμως, όταν έχουμε 1980 προϊόντα από διάφορα κράτη στην Ευρώπη, χρησιμοποιούν μια ετικέτα η οποία δηλώνει δεν περιέχει φινικέλαιο, ε, αυτό προξενεί βλάβη. 650.000 νοικοκυριά στη χώρα μου βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στο φινικέλαιο. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι τεράστιο το πρόβλημα. Όμως έχουμε δεσμευθεί ε, υπέρ των στόχων της κλιματικής, ε, για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Έχουμε δεσμευθεί ε, στο ότι θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά με τις κατάλληλες επιστημονικές επιτροπές. Όχι άλλη αποψήλωση στα δάση μας. Έχουν μείνει εκεί και ουρακουτάνγκια και μαϊμούδες, ναι. Κάνουμε το ανθρωπίνος δυνατόν για να εξασφαλίσουμε πώς θα παραμείνουν στη θέση τους και θα είναι τμήμα της χλωρίδας και της πανίδας. Οπότε είμαστε ανοιχτοί και στον ανταγωνισμό, αυτό σημαίνει εμπόριο. Όμως, ε, σας παρακαλούμε, ο ανταγωνισμός αυτός να οδηγεί σε δίκαιο εμπόριο, όχι μόνο σε ελεύθερο εμπόριο για μικρές α, ε, χώρες όπως η Μαλαισία. Τώρα, έχουν απαγγελθεί καταγυρίες σε πολύ κόσμο και αντιμετωπίζουν 35-40 ε, για παράδειγμα ε, για το θέμα αυτό, ε, για τα, την οικονομική διαφθορά. Για την Goldman Sachs είναι πιο ευαίσθητο, δεν θέλω να σχολιάσω. Θέλουμε εμείς να σεβαστούμε το κράτος δικαίου, οπότε αφήσουμε τα δικαστήρια να κάνουν τη δουλειά τους. Για την Κίνα οι εμπορικές μας σχέσεις είναι καλές, παρόλο που θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε κάποια από τα project τα οποία ενέκρινε η προηγούμενη διοίκηση. Το πρόβλημα με την Κίνα είναι ότι ακόμα και όταν ε, κοιμόμαστε ανησυχούμε για την Κίνα και όταν είμαστε ξύπνοι ανησυχούμε ακόμα περισσότερο. Είναι τεράστια χώρα, η παρουσία της είναι πολύ έντονη και θεωρούν πως όλη η θάλασσα της, η, της Νοτιού είναι δική τους. Ναι, όντως, και φέρει το όνομα αυτό, η θάλασσα της Νοτιού Κίνας, South China Sea. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά ελπίζω πως δεν θα κάνει το ίδιο και η Ινδία, γιατί τότε θα ζητήσει, ε, θα ε, κηρύξει μάλλον πως της ανήκει ο Ινδικός ωκεανός. Ξέρετε πως η Κίνα έχει ζητήσει να κάνει η ίδια την οριοθέτηση και η οριαθέτηση με, ε, που έχει κάνει μπαίνει μέσα στα δικά μας έδαφ, ε, ε, ε, ε, χωρικά ύδατα και πολλές φορές στέλνει ε, ακτεωρούς, που είναι μεγαλύτερος από το δικό μας ναυτικό σε μέγεθος. Οπότε καταλαβαίνετε πως τα θέματα είναι δύσκολα. Ακόμα δεν είχαμε κανένα επεισόδιο, αλλά ζητώ από τις Διεθνείς Επιτροπές και από την ΑΖΕΑΝ η θάλασσα αυτή να παραμείνει ελεύθερη από οποιασδήποτε ε, προσπάθει στρατικοποίηση. Εμείς ε, έχουμε υπογράψει την UNCLOS, που είναι η σχετική ε, σύμβαση του ΟΗΕ για το θαλάσσιο δίκαιο, έτσι ώστε να υπάρχει ελεύθερη διέλευση για όλα τα πλοία, αλλά δεν θέλουμε καμία περίπτωση όπου πολεμικά πλοία θα είναι παρόντα. Ήδη αντιμετωπίσαμε κάποιες μικροεντάσεις το Σεπτέμβριο. Δύο πολεμικά πλοία ε, βρέθηκαν σε μία απόσταση 40 περίπου μέτρων. Ξέρετε, για πολεμικό πλοίο το 40 μέτρα δεν είναι ε, καλή εξέλιξη και σε περίπτωση σύγκρουσης θα είχαμε πρόβλημα. Η ΑΖΕΑΝ εργάζεται στο θέμα αυτό με την Κίνα και έχουμε ήδη παρουσιάσει ένα ε, ενιαίο κείμενο, έτσι το ονομάζουμε, για την ε, συμπεριφορά που θα πρέπει να ακολουθούμε και αυτό ελπίζουμε σε δύο χρόνια να είναι έτοιμο έτσι ώστε να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της ε, Κίνας, την παρουσία της Κίνας στην θάλασσα της Νοτιοκίνας. Τώρα, εκδημοκρατισμός, ναι, Άλλο είναι να κερδίζει κανείς εκλογές και άλλο είναι να κάνει μεταρρυθμίσεις, αλλά γνωρίζουμε πως πάντα υπάρχουν θέματα τα οποία ε, μπορούν να εκτροχιάσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και θα πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί. Πιστεύουμε πως η νέα μας κυβέρνηση είναι σαφέστατα δεσμευμένη υπέρ της ε, συμμόρφωσης και του σεβασμού της δημοκρατίας ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Σας ευχαριστώ. Your Excellency Minister. Εξοχότατε. Σας ευχαριστούμε που ήρθαμε ευχαριστούμε για το χρόνο που μας αφιερώσατε για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με τα μέλη της Επιτροπής των Εξωτερικών. Ε, έπεται συνάντηση με τη Φεντερίκα Μοντερίνα από ό,τι γνωρίζω. Την είπατε εκπρόσωπο. Δώστε τις τα χαιρετίσματά μας. Καλή επιτυχία και στην κυβέρνηση και στη χώρα σας.